σημερινή συνεδρίαση. Επόμενη, ε, ξαναξεκινάει η συνεδρίαση αύριο στις 8.30. Έχετε την ατζέντα και μπορείτε να την βρείτε και στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρα στη συνεδρίαση.